Okay, members, if uh, Λοιπόν, παρακαλώ, αν θέλετε καθίστε να ηρεμήστε για να δούμε αν έχετε κάτι όλοι. Έχετε το κατάλογο ψηφοφορίας. Καταρχήν, η αθέτηση της σημερινής διάταξης δεν βλέπω να ζητά κανείς κάποια αλλαγή, οπότε θεωρώ πως συγκρίνεται και τώρα Έχουμε τις ανακοινώσεις της Πρόεδρου που αφορούν αποκλειστικό στους οικονομικούς διαλόγους, δηλαδή το διάλογο που κάνουμε με τους Υπουργούς Οικονομικών εδώ. Αύριο θα έχουμε έναν οικονομικό διάλογο λοιπόν με τον Ισπανό Υπουργό Οικονομικών ε, και όσον αφορά τη Γαλλία, στις 30 ε, Ιανουαρίου σας ενημερώνω ότι ο οικονομικός διάλογος αναβλήθηκε για δεύτερη φορά και ότι έχουμε ορίσει την 13η Φεβρουαρίου ως νέα ημερομηνία. Εν τω μεταξύ η γραμματεία της ΕΚΟΝ ενημερώθηκε ότι λόγω μιας άλλης απρόβλεπτης εκδήλωσης ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και Μοσκοβισή δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις συνεδρίες της ΕΚΟΝ στις 13 Φεβρουαρίου. Η τρίτη φορά που αναβάλλεται ο οικονομικός διάλογος. Εγώ θα έρθω σε επαφή με τον Υπουργό για να προγραμματίσω ξανά άλλη επαφή. Ελπίζω όχι πολύ ε, αργά. Όπως γνωρίζετε δεν μπορώ να υποχρεώσω έναν Υπουργό να έρθει, αλλά νομίζω πως δεν δίνει πολύ καλή εικόνα όταν αναβάλει για τρίτη φορά και φαίνεται σαν να φοβάται ή σαν να έχει κάτι να κρύψει. Και σίγουρα δεν μας εμπνέει εμπιστοσύνη. Ναι, καταλαβαίνω τις κυβερνητικές προτεραιότητες, αλλά ο οικονομικός διάλογος νομίζω πως είναι επίσης ένα πολύ χρήσιμος ε, μηχανισμός, όπως ε, άλλωστε ανακάλυψαν και διάφοροι Υπουργοί Οικονομικών, ώστε να εξηγήσουν ακριβώς ποια είναι τα προβλήματά τους και δεν, θεωρούν, και δεν βρίσκουν απαραίτητο εχθρικό ακροατήριο, αντίθετα μπορεί να τους βοηθήσει και όχι να τους βρίσκει ε, αντίπαλους. Όσον αφορά το Λουξεμβούργο έχουν υπάρξει καθυστερήσεις ε, στη διοργάνωση αυτού του οικονομικού διαλόγου λόγω της αλλαγής κυβέρνησης μετά από τον διορισμό του Δεκεμβρίου του κύριου Πιέρ Ομέγκο ως Υπουργό Οικονομικών και ελπίζω πως αυτό, αυτή η συνάντηση θα διοργανωθεί σύντομα. Και τέλος όσον αφορά την Πορτογαλία έχουμε επίσης ε, αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες και πάλι λόγω του ότι υπήρξε αλλαγή υπουργού Εν τω μεταξύ, μια αντιπροσωπεία τη ΕΚΟΝ ε, συνάντησε τον νέο Υπουργό στη Λισαβόνα στο πλαίσιο της έκθεσης ε, για τις δραστηριότητες της Τρόικα και θα συζητήσω το θέμα με τους συντονιστέ για το κατά πόσο θέλουν ε, να γίνει οικονομικός διάλογος αφού έγινε επαφή μέσω στο πλαίσιο της Τρόικα. Γενικότερα να πω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα μέσα και τα εργαλεία τα οποία έχουν υιοθετηθεί υπό το εξαπλό πακέτο και υπό το διπλό πακέτο χρησιμοποιούνται ε, αποτελεσματικά ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική συζήτηση στην Ευρώπη για αυτά τα σημαντικά θέματα. Και μάλιστα δεν μπορούμε να επιμένουμε για να κάνουμε εκθέσεις για την Τρόικα και μετά να θέλουμε και να μην εφαρμόζουμε τις εξουσίες που αποκτήσαμε μέχρι του εξαπλού και του διπλού πακέτου. Ακόμα και αν δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Οι οικονομικοί διάλογοι θα πρέπει να συζητίζονται, συνεχίζονται και όπως είπα πολύ συχνά βοηθούν και ε, πολλές φορές είναι και εξαιρετικά ε, λαμπερή και εντυπωσιακή γιατί μας έδωσε και κάποιες πληροφορίες για το πώς θεωρεί εκείνος ότι πρέπει να εργαζόμαστε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, πράγμα το οποίο θεώρησα ως αποκάλυψη εγώ προσωπικά. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία για την έκθεση περί ανταγωνισμού του Ανδρέα Σβάμπας. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Μάλιστα. Ζαν Πολ. Ναι, Πρόεδρε, εγώ ευχαριστώ. Ήθελα μόνο μια τεχνική ανακοίνωση να κάνω. Ζητώ από του συναδέλφου του ΕΛΚΑ να ακολουθούν το φίλο Αντρέα Σβάμπ κατ' εξαίρεση. Δεν είναι ο συντονιστή, αλλά ο Αντρέα που θα κάνει τι υποδείξει για την ψηφοφορία. Παρακαλώ λοιπόν να τον κοιτάτε στη διάρκεια τη ψηφοφορία. Okay, Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. ΕΛΚ, ο Αντρέα είναι εκεί για του ε, βουλευτές του ΕΛΚ, ο Αντρέα κάθεται εκεί. Λοιπόν, δοκιμή. Να Πατήσετε παρακαλώ τα κομβία. Μήπω μήπως έχει ε, ξεχάσει κανένα την κάρτα του. Περβάνς, μείον μια κάρτα. Έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚΑ. Δύο παραπάνω από το ΕΛΚΑ. Περβάνω, μήπως θα σου στείλει κανείς, θα σου φέρει κανείς την κάρτα σου, όχι. Οπότε θα πρέπει να μετράμε τους σοσιαλιστές κάθε φορά. Λυπούμε, αλλά... Well, we just need to count now. Ναι, εντάξει, να μετρήσουμε τώρα πόσοι ψηφίζουν. Παρακαλώ, μπορείτε να σηκώσετε όλοι οι σοσιαλιστές τα χέρια σας για να δούμε πόσοι είστε παρόντες. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 13. 13. How many supposed to have? Okay. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε ok με τα νούμερα. 13 είναι οι σοσιαλιστές. Προσθέτουμε λοιπόν την περβάνωση. Κανείς άλλος? Όχι. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Τροπολογία 99. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Εντάξει, να ελέγξουμε τη 17. «27 κατά 19 υπέρ, οπότε ε, απορρίπτεται όντως. Συμβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 καταπίπτει. Συμβιβαστική R, υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά αυτή τη συμβιβαστική, η R. One more to add in in favor. voted and that's rejected. Ψηφίσετε όλοι, απορρίπτεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή απορρίπτεται, νομίζω. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 137. Νομίζω πως είναι η ίδια πλειοψηφία. Thereof. Nobody's voted. That's one more in favour, but it's 23, uh, 23 γιατί έχουμε έναν ακόμα υπέρ, άρα απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο απορρίπτεται. Να ελέγξουμε και πάλι όμως. Oh, that's, that's Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε την 117, ούτε την 119 και ούτε τις υπόλοιπες μέχρι την 122, διότι είναι ψήφος για τους ορισμούς 106. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά νομίζω πως είναι η ίδια, το ίδιο αποτέλεσμα τέλος πληροφορίας ένας ακόμα υπέρ και απορρίπτεται 108 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14. Ελέγχουμε για την 110 πρώτα. Ναι, τη δική μου. Α, εγκρίνεται. Μπράβο που το έλεγξα. Σημαίνει ότι δεν είμαι προκατελημένη, έτσι. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. say definition there. Γιατί λέει εδώ ορισμοί. Λέει ότι ο ορισμός θα επικρατήσει. Yes, I think everything on collective redress has been rejected so far. But we can vote. This means that... Okay, so any bits that are definition... Εκεί που υπάρχουν λοιπόν ορισμοί, το κομμάτι του ορισμού επικρατεί, αλλά το υπόλοιπο επί της ουσίας ψηφίζουμε. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. 22 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εδώ έχουμε διαφορετικές, διαφορετικά νούμερα, το ελέγχουμε. Καταπίπτει γιατί είναι 23-23. 23 υπέρ, 22 κατά, αλλά η υπερβάση είναι κατά, οπότε απορρίπτεται. 116, all those in... υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω και αυτή απορρίπτεται. απορρίπτεται. Ήμκο 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τώρα στο 4, περνάμε στην 126. 126. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξω την 126. Everybody's voted and that's carried. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι, ήταν σαφέ νομίζω. Περνάμε στο συμβιβαστική β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 133 υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε, 133 Εγκρίνεται. Πάμε στην 25. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 26. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Συμβιβαστική C. Καταρχήν υπάρχει μια προφορική τροπολογία από την Άλτη και τους πράσινους. Ε, θα ψηφίσουμε λοιπόν πρώτα επί του κειμένου συμπεριλαμβανομένης της προφορικής τροπολογίας και αν αυτό καταπέσει τότε θα ξαναψηφίσουμε χωρίς την προφορική. Με την προφορική ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είδα. Καλύτερα ηλεκτρονικά να ελέγξουμε. Απορρίπτεται εντελώς. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ψηφίσουμε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται I can find it it's on page it's on page 11 in CA although Συμβιβαστική CA, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. CA. Συμβιβαστική CA. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική CB. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Jury 23. In favor. Jury 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 45. Yes, indeed, that is carried. Uh, and then 100 so falls. Ωραία λοιπόν, εγκρίνεται και πάμε στην επόμενη σελίδα που είναι η 46. Τροπολογία 46, ποιοι είναι υπέρ. 46, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 177, υπέρ. Κατά. Αποχές, έχουμε ηλεκτρονικά για την 177. Δεν είναι εύκολο να δει κανεί αν εγκρίνεται ή αν απορρίπτεται. Λοιπόν, εγκρίνεται αυτή. 24 προς 22. 4, No. 178. 178. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 182. 23-23, άρα καταπίπτει. 32 ε, ήταν, συγγνώμη. 180 υπέρ. Κατά αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Διότι έχουμε διάφορες ενδιαφέροντες, διάφορους ενδιαφέροντες συνδυασμούς. Ένας ακόμη. Τέλος ψηφοφορίας. Και καταπίπτει. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, μάλλον καταπίπτει, αλλά να το ελέγξουμε. Καταπίπτει. Ήμκο 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Πάλι στην κόψη είναι. Εγκρίνεται, δεν εγκρίναμε και κάτι, ωραία. 182 υπέρ. Κατά. Εποχές. Ε, ελέγχουμε και την 182. Εγκρίνεται. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, έχει καταπέσει ούτως ή άλλως. Θα ελέγξω την 183. Απορρίπτεται. 48. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Στη 49 πρέπει να ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές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 ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Μας έμενε λοιπόν μόνο το πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής D. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει κάτι άλλο να ψηφίσουμε, όχι. Πάμε στη συμβιβαστική E. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 55, τροπολογία 55 υπέρ. κατά. Αποχές απερίφθει αλλά επαληθεύουμε την 55. Απερίφθη. 198 υπέρ 198 κατά. Αποχές επαληθεύω την 198. Απερίφθη. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική F. Προφορική τροπολογία πρώτα. Προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε είναι διαφορετικός ο συνδυασμός της ε, ψήφους. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε σε τμήματα. Πρέπει να γίνει σε τμήματα πάλι μετά την προφορική τροπολογία. Πράσινη τι λέτε. γιατί αλλάξαμε το passing on το κομμάτι αυτό. Άρα, από ό,τι βλέπω εγώ, θα χρειάζεται σε έτσι δεν είναι. Καλώς. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβαστική G. Ζήτα. Υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε παρακαλώ συμβαστική G «23 υπέρ, 23 κατά» λέει η πρόεδρος, άρα απορρίφθη. Απορρίπτεται. 205 ε, τώρα υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 206 υπέρ Γιατί να καταπίπτει αφού λέτε ότι καταπίπτει, αν καταπίπτει. Ε, ο εγκέφαλος μου δεν αντιλαμβάνεται πώς μπορεί να καταπέσει μια ανθρωπολογία και καταπίπτοντας να κάνει μια άλλη να καταπέσει. Αν και έχει ξανασυμβεί. Εν πάση περιπτώσει δεν καταπίπτει είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς να ξέρει ποτέ. 206 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα το επαληθεύσουμε. Πρέπει να ψηφίσει ακόμη ένας. Εγκρίνεται λοιπόν. Με σημαντική πλειοψηφία. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές την επαληθεύουμε παρακαλώ 207 και στο συγγνώμη για τις επαληθεύσεις. Αλλά είναι πολύ ακατάστατη η ψηφοφορία. Δύο ακόμα συναδελφοί δεν έχουν ψηφίσει. Παρακαλώ. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23-23 εάν είναι και κατά. Άρα απερίφθη. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 33 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 209 έχει απορριφθεί. 210 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 212 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε 212. Μια νέα ακόμα ένας να ψηφίσει παρακαλώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 61 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 της Επιτροπής ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά... Ήταν διαφορετικός ο συσχετισμός των ψήφων. Απερίφθη. Έχουμε μία κάρτα μήπως παραπανήσια. Ή δεν δουλεύει. Όχι, είχατε πει ότι ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε από το ΕΛΚ. Ήθελα να επαληθεύσω λοιπόν. Τι γίνεται. Όχι, έχει απορριφθεί. Κλείνουμε αυτή την ψηφοφορία. Ξέρετε, αν εμφανιστούν πολλές κάρτες, περισσότερες από ό,τι πρέπει, βγαίνει ένα μήνυμα από το μηχάνημα. Συμβαστική H, λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική Y, I, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές Α, όχι, ξαναρχίζω. Πρώτο τμήμα της J, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, κατά, αποχές, επαληθεύουμε για το δεύτερο τμήμα. Ψήφισαν όλοι, εγκρίνεται. 226. Τροπολογία 226 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 227 και 48 της Επιτροπής Ιστορικής Αγοράς υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε. Δεν ε, προχωράει πολύ γρήγορα το μηχάνημα σήμερα. Περίφθη. 228 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε την 67, αλλά νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Ακόμη ένας. που έχουν ψηφίσει. Πέρας προφορίας εγκρίνεται. Ένα τη ΣΥΜΚΟ υπέρ. Είναι συμπαθήνα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την τροπολογία παριθμών 1 της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Ψήφισαν όλοι. Απερίφθη. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές επελθεύουμε την 68, αν και νομίζω ότι έχει και αυτή απορριφθεί. Απερίφθη. Με μία ψηφοδιαφορά. Δύο της ΕΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη επολυθεύουμε την 71 ψήφισαν όλοι 26 κατά 27 απερίφθη 72 υπέρ Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 72. Επαληθεύουμε την 72. Απερίφθη. Ακόμη και αν είναι υπέρ, απερίφθη. Η τρία της ΕΜΚΟ υπέρ, κατά. Αποχές. Απερίφθη. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές Απερίφθη. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν τη 2. Δύο ακόμα μένει να ψηφίσουν. Πέρας. Απερίφθη. 26 κατά δηλαδή. Η 73 παρακαλώ. Να κύριε Σφάπ. Χωρίς μικρόφωνο. Ήταν πολύ στενά τα περιθώρια στην ψηφοφορία G για τη συμβαστική J. Μια και, μια και επιτρέψα στην κυρία Σαϊά να ξαναψηφίσει και ήταν τόσο στενά τα περιθώρια και νομίζω ότι είχε αλλάξει. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Όχι, λέει η πρόεδρο, με τι συνθήκε που είχε η αίθουσα την ώρα που ήταν η ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι α, ήρθε κάποιο και ξαναψηφίζουμε. Δεν, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Για τότε θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, να ξανακάνουμε ολόκληρη την ψηφοφορία, γιατί μπορεί να φτάσει κάποιος άλλος συνάδελφος. Ένα λεπτό. Ήμασταν στη διάρκεια της ψηφοφορίας της συμβαστικής και κάποιος ρώτησε πώς πήγε η ψηφοφορία και εγώ είπα να επανέλθω γιατί δεν είχα επαληθεύσει. Όσο γίνεται η ψηφοφορία μιας συγκεκριμένης τροπολογίας επαληθεύω. Αλλά δεν θα κάνω ε, πέντε βήματα πίσω όταν βλέπω ότι αλλάζουν οι κάρτες, μπαίνουν και βγαίνουν συνάδελφοι. Διαδικαστικά δεν είναι σωστό αυτό, γιατί προσπαθώ να είμαστε δυνατόν πιο ισοδίκαιοι και να επαληθεύω στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αλλά αυτό πια παραπάει. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 73. Ψηφίστε παρακαλώ. Απορρίφθηκε. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ίδια πλειοψηφία. 77 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 ήμκο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Α, όχι, συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρος. Εγκρίθηκε, σωστά. Τροπολογία 80 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. Εγκρίθηκε. 82 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα για την 83. Ψηφίστε παρακαλώ. Άλλο ένα Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδια πλειοψηφία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Τζούρι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Εμκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 8 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Απορρίφθηκε. 9. Υπέρ. Του συγητή, έτσι. Ναι, του συγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την εννέα, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίθηκε. Ήμκο εννέα. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 92 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 92 παρακαλώ. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 τζούρι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Εγκρίθηκε. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 14 ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 93 καταπίπτει. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά, αποχές, θα ελέγξουμε 15, ψηφίστε. Εγκρίθηκε. Ίμπκο, όχι καταπίπτει, 94 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε και εδώ. Τι να κάνω. Πέρα τη ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 16 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για το πρώτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα, αν και δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα. Καταπίπτει νομίζω και δεν έχει νόημα από μόνο του. Οπότε πάμε στην τροπολογία 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 97. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Απορρίπτεται νομίζω. Εγκρίθηκε. Συνεπώς. Θέλετε διάλειμμα. Για να ξέρουμε τι κάνουμε. Όχι. Καλά. Συνεχίζουμε. Τότε ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το τροποποιημένο κείμενο παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές. Ε, ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου τώρα. Πάλι ηλεκτρονικά ψηφίστε. Α, μία ψήφοι πέρα αυτή τη φορά, δύο κατά και 4 αποχές. Κύριε Σιγητά, θέλετε να ξεκινήσετε διαπραγματεύσεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα σας κρατήσω. Ευχαριστώ όλους και ηγητές από τις άλλες ομάδες. Μπορούσαμε σε πολύ στο χρονικό διάστημα να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις και πολλά σημεία. Πρέπει να πω ότι καθοριστικής σημασίας ε, σημεία, τροπολογίες απερίφθησαν με ψήφους μόλις 23 προς 23. Δεν είναι αυτό καλή γερή βάση για διαπραγματεύσεις, ε, για αναζήτηση δηλαδή πολιτικών βουλήσεων. Ε, γι' αυτό παρακαλώ να ε, το λάβουμε υπόψη και να μου χορηγηθεί βέβαια η εντολή για την πραγματεύση. Πρόεδρο, ψηφίζουμε τότε για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Α, κύριε Λάγκε, θέλετε κάτι? Με τόσες ψηφοφορίε οι οποίες εξαρτήθηκαν από μία μόνο ψήφο και τόσο σημαντικής, ε, τόσο μεγάλη σημασία ψηφοφορίες, νομίζω ότι το θέμα πρέπει να φτάσει στην Ολομέλεια για να κρυθεί εάν θεωρεί ο εισηγητής ε, ότι είναι σκοπό. Αν και νομίζω ότι δεν του διευκολύνω το έργο με αυτό που λέω. Συμφωνώ με τον Λάγκε. Προσωπικά μιλάω. Δεν νομίζω ότι μας συμφέρει να πάμε σε τριμερή διάλογο με ψηφοφορία που κρίθηκε από μία ψήφο, καμιά φορά στην τύχη δεν είναι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να πάμε πρώτα στην Ολομέλεια. Για μένα είναι ο μόνος ορθός τρόπος για να χειριστούμε ένα τέτοιο ζήτημα. Πρόεδρος, αντιλαμβάνομαι τα σχόλια. Άρα μπορούμε να ψηφίσουμε την απόφαση να μπούμε ή όχι σε διαπραγματεύσεις. Χρειαζόμαστε 26 ψήφους υπέρ προκειμένου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Πέρας της ψηφοφορίας. 33 ψήφοι υπέρ και 12 κατά. Καμία αποχή. Συνεπώς η διαπραγματευτική ομάδα θα είναι πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, εισηγητής και σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ. And for those who are anxious, the next meeting... Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα την 3η 28 Ιανουαρίου στις 4 το απόγευμα.